ευρώ το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια του EP Justa έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, η απόδοση ποινική δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταλή. Έχουμε ε, επτά ψηφίσματα στο τέλος της συζητήσεως, τα οποία θα ψηφιστούν στο τέλος. Μετά την επόμενη συζήτηση, ακολουθεί τώρα η συζήτηση της κατάστασης των εθνοτικών μειονοτήτων στο Ιράν και από τους συντάκτες ξεκινάει ο κύριος Πάσκα ε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, στο Ιράν οι πολιτικοί ε, ακτιβιστές έχουν πρόβλημα για την αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τις ε, θρησκευτικές, ε, εθνοτικές και άλλες μειονότητες. Απευθύνουμε έκκληση στις Ιρανικές Αρχές προκειμένου να επιτρέψουν στις μειονότητες να χρησιμοποιούν την γλώσσα τους στην επικοινωνία μεταξύ τους και να μπορέσουν ελεύθερα να ασκούν τη θρησκευτική τους λατρεία, να σταματήσουν οι διακριτικές μεταρρυθμίσεις και οι διώξει των μειονοτήτων για θρησκευτικούς, εθνοτικούς, γλωσσικούς ή άλλους γνώμους, λόγους. Η, δυστυχώς είναι πολύ αλαζονική η στάση της Ιρανικής κυβέρνησης. θα πρέπει να έχει υπόψη της, η κυβέρνηση αυτή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί την κατάσταση εκ του σύνεγγυ και κάποιες ειδήσεις θα ζητήσει ευθύνες για αυτή την αλαζονική πολιτική εις βάρος των μειονοτήτων. Ευχαριστώ τον κύριο Πάσκα, ο κύριο Σταβάρες για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι ανησυχητική κατάσταση στο Ιράν, ε, η κατάσταση των μειονοτήτων. Είναι πολύ σοβαρή και μάλιστα συνεχώς επιδεινώνεται. Επίσης η πολιτική κατάσταση στο Ιράν ούτως ή άλλως είναι περίπλοκη ακόμη και για την πλειοψηφία των Περσών Ιρανών που και αυτοί δεν μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματα Το Γνωρίζουμε ότι στις εκλογές έγινε νοθεία. Είχαμε απαγωγές εθνικό, εθνοτικών μειονοτήτων στις, ε, και μάλιστα οι φυλακισμένοι εθνοτικών μειονοτήτων ε, ε, λαμβάνουν πολύ χειρότερη μεταχείριση από τους υπόλοιπους Ιρανούς. Το, το σύστημα της δικαιοσύνης επίσης προβαίνει σε διακριτικές μεταχείρισεις εις βάρος των εθνοτικών μειονοτήτων. Η κατάσταση των γυναικών εθνοτικών μειονοτήτων είναι πολύ χειρότερη από των, των υπόλοιπων ε, γυναικών. Η κατάσταση σχολεία είναι πολύ χειρότερη. Πολύ ζωφερό αυτό το πλαίσιο και το τοπίο και πολύ ανησυχητικό. Ε, δυστυχώς ε, συνεχίζεται και αυξάνεται και η χρήση της θανατικής καταδίκης, της θανατικής ποινής στο Ιράν. Ακόμη και για εγκλήματα σεξουαλικού προσανατολισμού και μάλιστα εκτελούνται ακόμη και νέοι. Απευθύνουμε έκκληση λοιπόν στην Ιρανική κυβέρνηση για να θέσει επιτέλους τέρμα στις ε, διακριτικές αυτές μεταχειρήσεις και για να τροποποιήσει τη στάση της απέναντι στις μειονότητες. Βέβαια δεν έχουμε και πολλές ελπίδες ότι θα μας ακούσει και θα αλλάξει τη στάση της Ιρανική κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να σκεφτεί αυτό που κάνει. Ε, δυστυχώς ε, με τις ε, πρακτικές αυτές ε, διχάζει τον εθνοτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό ιστό του Ιράν και σπέρνει ε, τη, τους σπόρους της διχόνοιας και του μίσους για το μέλλον. Θα πρέπει το Ιράν να αναφροντίσει ε, να δημιουργηθεί μια ομόνια μεταξύ των εθνωτικών μειονοτήτων και ίσως με τέτοια συνεργασία μπορεί κάποια στιγμή να ανατραπεί και η κυβέρνηση. Ευχαριστώ και για ένα λεπτό τώρα κυρία Ντεκάιζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ο λαός του Ιράν αποτελείται μόνο κατά το ίμιση από Πέρσες. Οι υπόλοιποι είναι διαφορετικές εθνότητες και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών κατά των φιλετικών διακρίσεων έχει ε, ήδη σημειώσει τις, ε, ε, τις διακρίσεις κατά πολλών εθνοτήτων, Τουρκμενών, Κούρδων, Αράβων. Υπάρχουν μία, υπάρχει μία μικρή ομάδα Αράβων Ουαζί οι οποίοι ε, ε, ε, διώκονται και κάθε Απρίλιο υπάρχουν διαδηλώσεις το 2011 φαίνεται ότι αυτές οι διαδηλώσεις οδήγησαν σε 12 θα, 15 θανάτους και ορισμένους τραυματισμούς που αναφέρθηκαν στο facebook και τώρα υπάρχει ε, ένας ε, ε, ένα άτομο που σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν και 15 πρέπει να δικαστούν αλλά είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρώσουμε σωστές πληροφορίες παρόλα αυτά πιστεύω πιστεύω ότι στο σημείο 3 το γεγονός και μόνον ότι ονομάζουμε τους κυρίους αυτούς ε, και ζητώντας να δικαστούν δίκαια ε, είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ. Κυρία Ντεκάιζερ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Σάκε για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Είναι γεγονός ότι οι Ιρανοί ζουν ε, σε ένα κράτος βίας κάθε μέρα ε, ε, και βεβαίω αυτό το στοιχείο δεν θα πρέπει να ξεχαστεί στην διαπραγμάτευση ε, με, που αφορά την πυρηνική ενέργεια. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ε, στρατηγικής σημασίας και δεν μπορούν να μπουν σε μια ζυγαριά ε, μαζί με το πυρηνικό πρόγραμμα. Αυτή τη στιγμή υφίστανται μεγάλη διακριτική μεταχείριση οι μειονότητες και οι διαφορετικές εθνότητες. Γνωρίζουμε ότι το Ιρανικό καθεστώς είναι γνωστό, είναι διαβόητο για την βία με την οποία αντιμετωπίζει τους ε, πολίτες, τους βασανιστήρια, κρατήσεις, ε, θανατώσεις κλπ. Θα πρέπει να ζητήσουμε από τις ε, Ιρανικές αρχές να εφαρμόσουν τα όσα προβλέπει το δικό τους σύστημα Σύνταγμα, συγγνώμη, ε, θα πρέπει ε, να ε, δώσουν τη δυνατότητα σε όλες τις εθνότητες να ζήσουν ειρηνικά. Θα πρέπει να ελευθερώσουν όλους τους ακτιβιστές οι οποίοι έχουν συλληφθεί λόγω της δράσης τους για την προστασία των μειονοτήτων. Θα πρέπει ο καθένας να μπορεί να μιλάει τη γλώσσα του, να έχει εκπαίδευση στη γλώσσα του και να ζει ειρηνικά στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Κόρολα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ και δύο χρόνια ένας ε, γνωστός ε, δάσκαλος ε, ιρανοκουρδικής καταγωγής δολοφονήθηκε. Ο ο δολοφόνος του καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση. Έχουμε επίσης και άλλες περιπτώσεις. Έχουμε περιπτώσεις όπου έχουν διωχθεί ε, άνθρωποι ε, λόγω ε, με την κατηγορία της αποστασίας, δηλαδή της απομάκρυνσης από το λόγο του Θεού. Οι Ιρανικές αρχές στην ουσία κάνουν ό,τι θέλουν. Στο Ιράν αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες ε, θρησκευτικές μειονότητες ε, μεταξύ των οποίων και οι Εβραίοι και οι ε, Χριστιανοί αλλά έχουμε και άλλες μη αναγνωρισμένες μειονότητες όπως είναι οι αχβαζ η Μπαλούχ κτλ. Υπάρχουν λοιπόν μία σειρά ανθρώπων οι οποίοι δεν μπορούν ούτε να μιλήσουν τη γλώσσα τους ούτε να ασκήσουν τα θρησκευτικά τους δικαιώματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Βερζιά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πριν από μερικές μέρες ε, οι Κούρδοι του ε, Ιράν ε, είχαν μια εκδήλωση για, το θάνατο του Μεχμίτ Τζαλία, ο οποίος πέθανε μετά από τέσσερα χρόνια στην φυλακή και βεβαίως όλοι ε, αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν τελικά στη φυλακή εκατηγορούνται ε, για κακή χρήση του ονόματος του Θεού. Ε, ξέρουμε ότι οι συλλήψεις είναι πολλές και οι συλλήψεις των Κούρδων, των Ιρανών Κούρδων είναι πολλές και δεν είναι οι μόνοι και οι Αζέρι και οι Άραβες και οι Μπαλόχ και οι Αχβάζ έχουν υποστεί μεγάλες διωγμές. Επίσης δεν είναι καλό να είναι κανείς γυναίκα στο Ιράν, δεν είναι καλό να ζει στο Ιράν, ε, δεν ε, είναι ε, δυνατόν να δεχόμαστε μια κατάσταση όπου θανατώνονται όλο και περισσότεροι άνθρωποι και όλο και περισσότερα παιδιά μεταξύ αυτών. Και εμεί τι κάνουμε, μιλάμε εδώ στο Κοινοβούλιο, ήρεμα και ωραία, περιμένοντας μέχρι την επόμενη φορά που θα έχουμε κάποιε νέε παραβιάσεις. Και βεβαίω οι ιρανικέ αρχέ επιτρέψτε μου να πω, ότι δεν νοιάζονται καθόλου. Η κυρία ε, Λέιλα Ζάνα, ε, παρόλα αυτά, ε, είναι, ήταν στη φυλακή τόσα χρόνια, έστω και αν ήταν βραβείο Ζαχάροφ. Το ίδιο γίνεται και με, τους, με το Ιράν. Ο κύριος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι πραγματικά λυπηρό που το Ιράν, μια χώρα με πολύ όμορφο πολιτισμό, μακροχρόνια παράδοση, τεράστια πανέμορφη χώρα ε, διακυβερνάται από μια κυβέρνηση που δεν ε, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, προβαίνει στη διακριτική μεταχείριση των μειονοτήτων, καταπιέζει τον ίδιο τον πληθυσμό και έχει και ε, βλέψεις για πυρηνικά όπλα. Βλέπουμε ότι γίνονται διώξεις χριστιανών αλλά και άλλων εθνοτικών μειονοτήτων στη χώρα αυτή. Φυσικά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Βέβαια δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Είμαστε σχετικά ανήμποροι γιατί οι Ιρανικές αρχές έχουν ανοσία απέναντι στις επικρίσεις και στις μομφές. αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να διατρανώσουμε τη διαφωνία μας με την κατάσταση αυτή και την συμπεριφορά αυτή που θα πρέπει να τη στυλιτεύσουμε. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε τη δραστηριότητα ε, της Ιρανικής Αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι αυτή, αν άλλο, είναι μια προσπάθεια να ασκήσουμε πίεση στις Ιρανικές Αρχές. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Βοητσεχόφσκι. Ε, ευχαριστώ κύριε Βοησικόφση. Αυτή ήταν η συντάξει και τώρα έχει το λόγο ο κύριος Πόισελτ για ένα λεπτό σαν πρώτος ομιλητής. Κύριε Πρόεδρε, το Ιράν εξετάζεται μονολυθικά σαν σιητική μονάδα. Είναι όμως ε, ένα πολυπληθυσμιακό κράτος το οποίο ε, έχει ε, χριστιανικές μειονότητες οι οποίες πάνε καλά όπως οι Αρμένοι, άλλοι όμως διώκονται όπως οι Ασσύριοι, οι χριστιανοί γι' αυτό και διάφοροι υποφέρουν και εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε το Ιράν σε όλη την ποικιλομορφία του να εξασφαλίσουμε ότι οι μειονότητες ε, θα προστατεύονται και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να ασχολόμαστε τακτικά με το Ιράν διότι πολλές φορές τα ίδια έγιναν με το Ανατολικό Μπλοκ και ε, βλέπουμε ότι κάποια στιγμή όταν θα είναι ελεύθερες ε, πολλές, ε, ε, πολλές κοινότητες θα μπορέσουν να συμβιώσουν στο Ιράν και να είναι οι εταίροι μας. Ευχαριστώ κύριε Πόσελ. Το λόγο έχει τώρα η κυρία Γιούλαντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν μας εκπλήσουν στο Ιράν διότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει ε, καταγραφεί και συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επανειλημμένο στο παρελθόν. Έχουμε ζητήσει από τις αρχές να καταργήσουν όλες τις ε, διακρίσεις και να επιτρέπουν την ελεύθερη ε, άσκηση θρησκειών και συγκεντρώσεων. Αλλά ξέρουμε ότι το ψήφισμα αυτό θα παραγνωριστεί όπως έγινε και στο παρελθόν. Παρόλα αυτά ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να προβεί σε συζητήσεις με το Ιράν ε, κατά τρόπον ώστε ε, να μπορέσει κανείς να στηρίξει μία ε, κατάλυση του φονταμεδεσταλιστικού καθεστρώτος και να υπάρξει μία εναλλακτική κατάσταση η οποία θα μπορέσει να επιταχυνθεί. Ευχαριστώ κυρία Όγιουλαντ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ιράν είναι μια χώρα που η διακυβέρνηση ασκείται με βία εις βάρος των πολιτικών αντιπάλων, εις βάρος εθνοτικών και θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα εις βάρος των χριστιανών που εδώ και χρόνια υφίστανται αυτές τις διώξεις και χάνουν τη ζωή τους για την πίστη τους. Δεν είναι εύκολο να είναι κανείς καθολικός στο Ιράν. Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει ρίζες στον χριστιανισμό θα πρέπει να ε, προστατεύσει τα δικαιώματα αυτών των μειονοτήτων γιατί το δικαίωμα στη θρησκεία είναι ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα του ανθρώπου. Δεν θα πρέπει για κανένα λόγο, είτε οικονομικό είτε πολιτικό, ε, να ανεχόμαστε αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Να απευθύνει έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει οποιαδήποτε προσπάθεια προκειμένου να προασπίσει τα δικαιώματα των χριστιανών στο Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκρόμπατσικ. Αυτό όσον αφορά τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σιλβέστρης το νομικό σύστημα, το δικαστικό μάλλον σύστημα ε, της Ιρανικής Δημοκρατίας ε, έχει ε, οδηγήσει, έχει καταδικάσει 600 ε, πολίτες σε 300, σε 300 χρόνια κράτηση. Στο Ιράν είναι πολλά τα εμπόδια για αυτόν που προσπαθεί να δώσει δικαιώματα στις μειονότητες γιατί δεν δίνει αυτή η Ιρανική Δημοκρατία την δυνατότητα στους ε, ανθρώπους που προέρχονται από μειονότητες οποιοδήποτε είδους ε, να ζήσουν ε, με σεβασμό των δικαιωμάτων τους. Βλέπουμε επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες αρνητικές τάσεις. Δηλαδή επιτείνεται η, πίεση των χριστιανικών και το τονίζω και δεν καταλαβαίνω δεν θέλουμε να το πούμε στα ψηφίσματά μας των χριστιανικών μειονοτήτων. Πιέζουν όλο και περισσότερο τις χριστιανικές μειονότητες. Επίσης αυτούς, ε, αυτοί που ε, ανήκουν σε θρησκευτικέ μειονότητες ε, θεωρούνται σίγουρα δεύτερης ποιότητας πολίτες και οπωσδήποτε σχεδόν παράνομοι. Ευχαριστώ. Τώρα ερχόμαστε στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ και σας ζητώ την κατανόησή σας γιατί σε αυτό το φλέγον θέμα έχουν ζητήσει το λόγο πάρα πολύ και δεν θα μπορέσω να τους καλύψω όλους. Ο, ο Σόνικ. Ε, ευχαριστώ. Εδώ και χρόνια βλέπουμε στο, ότι στο Ιράν καταπατώνται τα ε, δικαιώματα, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα πολιτιστικά των εθνοτικών, θρησκευτικών και άλλων μειονοτήτων. Καταπατούνται ε, και τα δικαιώματα που, χαρ, κατοχυρώνονται στο χάρτη ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, Παρ' όλα αυτά το, και επίσης το Ιράν είναι η χώρα που εφαρμόζει κατα, ε, ε καταξοχήν την θανατική ποινή, ακόμη και ε, εις βάρος ανθρώπων που δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλημα. Ε, είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση της σουνητικής ή της κουρδικής μειονότητας που κατηγορούνται πολλές φορές για κατασκοπία. Δημιουργείται ένα κλίμα εκφοβισμού, γίνονται μαζικές συλλήψεις. Θα πρέπει λοιπόν να κρούσουμε τον κόδωνα του κινδύνου για την καταστρατήγηση αυτή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν και να απευθύνουμε έγκληση προς το Ιράν να τηρηθεί το Σύνταγμα και να γίνουν οι απαραίτητε αλλαγές στον ποινικό κώδικα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα τα δικαιώματα των ε, θεωρητικών και άλλων μειονοτήτων. Επίσης, ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε τις επαφές ε, μέσω της αντιπροσωπείες που έχουμε για τη σχέση με το Ιράν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Σόνικ. Η κυρία Κροτού τώρα κρετού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να στείλουμε ένα ηχηρό και κατηγορηματικό μήνυμα προς τις Ιρανικές Αρχές ως προς την ανάγκη να παγώσουν πάρα αυτά οι θανατικές καταδίκες εις βάρος των μελών της αραβικής κοινότητας που κινδυνεύουν να εκτελεστούν ανα πάσα στιγμή. Οι άνθρωποι αυτοί αξίζουν μιας δίκης δίκης ε, και θα πρέπει ε, και οι οικογένειές τους να ανακουφιστούν. Επίσης θα πρέπει να σταματήσουν τα βασανιστήρια και ε, τα στρατόπεδα Κράτηση στα οποία επικρατούν απάνθρωπε συνθήκε. Θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τις ιρανικέ αρχές να καταργήσουν τη θανατική ποινή και να αναστείλουν τις διώξει των διαφόρων μειονοτήτων. επίση πιστεύω ότι θα πρέπει να εντείνουμε τις συνεργασίες με τον ΟΗΕ για τα θέματα αυτά. Ο κύριος Βλάσακ, για ένα λεπτό. Όταν ε, συζητούμε θέματα εθνοτικών μειοτήτων και τα δικαιώματα τους θα πρέπει ε, οπωσδήποτε ε, να αναφέρομαι και τα δικαιώματα των Ιρανών πολιτών ε, σε στρατόπεδο του Ιράκ που ζουν διαρκώς με καθεστώς φόβου και απειλής σε φρικτές υγειονομικές συνθήκες. Οι βαρόνοι Άστον γνωρίζει το ζήτημα αυτό και έχει ζητήσει άλλωστε να λυθεί αυτή η φλέγουσα κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Γεντζαγεύσκα για ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πολύ δύσκολη κατάσταση των μειονοτήτων στο Ιράν σχετίζεται άμεσα με την ε, έλλειψη της ανεξαθρησκείας στη χώρα αυτή και την έλλειψη ελευθερίας θρησκευτική ε, έκφρασης. Αναφέρθηκαν πολλά χαρακτηριστικά παραδείγματα δίωξη εθνοτικών ε, και θρησκευτικών μειονοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανών. Δεν θα επαναλάβω τα σχόλια αυτά. Θα ήθελα απλώς να πω ότι ε, εμένα προκαλούν μεγάλο πόνο οι απαγγελίες θανατικών ποινών για ανθρώπους που άλλαξαν πίστη, που απαρνήθηκαν το Ισλάμ. Αυτό αποτελεί κατάφορη παραβίαση του ανθρώπινου δικαιώματος της ελευθερίας θρησκευτικής πίστης. Τέτοιου είδους εκτελέσεις είναι απαράδεκτες και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνονται. Ευχαριστούμε κυρία Γιάννη Για το τέλος ε, της, κυρίας, ε, της διαδικασίας Κάτσου ο κύριος Κίνερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Ντεκάιζερ είχε δίκιο όταν είπε ότι δεν είναι μονοπολιτιστική κοινωνία το Ιράν παρόλο που είναι μία μουσουλμανική δημοκρατία. Όντως είναι πολύ επικίνδυνο να είναι κανείς εθνική ή θρησκευτική μειονότητα στο Ιράν αλλά πρέπει να υπάρχει γενική εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλες τις ε, εθνικές ε, ε, ε, σε όλες τις και σε όλες τις θρησκευτικές ομάδες. Αλλά βλέπουμε ότι αυτοί που έχουν προσιλητιστεί σε άλλες θρησκείες κινδυνεύουν και ίσως και περισσότερο από τις γνωστές μειονότητες. Ως εκ τούτου θα ήθελα να υπάρχει μία ευρία κάλυψη των μειονοτήτων, όχι μόνο των χριστιανών, να περιληφθούν στη δήλωση Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκίνερ. Έτσι ολοκληρώνεται η διαδικασία Catch the και στο τέλος θα λάβει το λόγο για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Επίτροπος Νταλή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Όπως υπόθηκε, το Ιράν είναι μοσαϊκό πολιτιστικό τουλάχιστον 40% του πληθυσμού ε, δεν είναι περσικής καταγωγής. Ε, πρόκειται για Αζέριους, ε, για Μπαλόχ, για Μπαχάης, για Τουρκμένους, Ασσύριους, Γεωργιανούς κτλ. Τοποθετούνται στην περιφέρεια κυρίως παρά τις ε, συνταγματικές διασφαλίσεις οι Ιρανοί οι οποίοι ανήκουν σε μειονότητες υφίστανται διακριτική μεταχείριση ε, που μπορεί να ε, σημαίνει ότι έχουν περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματά τους σε συγκεκριμένες παραβιάσεις ε, ε, καθώς επίσης ε, και δικάζονται χωρίς λόγο και καταδικάζονται συχνά σε θανατική ποινή. Επίσης συστηματικά τους αρνείται το δικαίωμα του συνέρχεστε και του μετακινήστε καθώς επίσης οπωσδήποτε δεν μπορούν να φτάσουν σε κάποιες κυβερνητικές θέσεις. Ε, στην, ε, στο Αζερμπαϊτζάν ε, καθώς επίσης και στο Χαουάζ βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα. Όλα αυτά έχουν ανησυχήσει τα Ηνωμένα Έθνη. Το ψήφισμα του Νοεμβρίου 2011 για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν το καταδεικνύει τα Ηνωμένα Έθνη ε, έχουν ε, ε, υπογραμμίσει διάφορες παραβιαστικές τακτικές και διακριτικές πρακτικές κατά των μειονοτήτων στο Ιράν και τις έχουν καταδικάσει πρέπει οπωσδήποτε να εγγυηθεί η κυβέρνηση τα δικαιώματα όλων των πολιτών του Ιράν ε, ε, εμείς προσπαθούμε να παρακολουθούμε όλες τις ε, περιπτώσεις διακριτικής μεταχείρισης που οφείλονται στο φύλλο, στον σεξουαλικό προσανατολισμό, στην εθνότητα ή στην θρησκεία χρησιμοποιήσαμε και χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία τα οποία έχουμε στην διάθεσή μας έτσι ώστε να ζητήσουμε από το Ιράν ε, να σταματήσει τις ε, διακριτικές ε, πρακτικές. Ε, και ε, ε, η ίδια η Βαρόνια Άστον και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γενικότερα έχουν επανειλημμένα αναφέρει ακόμα και με μονομένες περιπτώσεις στον Ιούνιο του 2011 ας πούμε στην Τεχεράνη απαγγέλθηκε κατηγορία θανατικής ποινής σε τέσσερις Κούρδους ε, και η Αντιπρόεδρος ε, ε, Άστον και σε αυτή την περίπτωση αλλά και σε άλλες παρόμοιες έχει εκδώσει ανακοινοθέντα καταδικάζοντας τις πρακτικές αυτές. Βεβαίως εμείς είμαστε ε, πάντα ανοιχτή ε, σε διάλογο ε, με την Ιρανική κυβέρνηση όσον αφορά την συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρ' όλα αυτά έχουν ληφθεί περιοριστικά μέτρα για 28 άτομα που βρίσκονται στον κατάλογο παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του Ιράν. Ευχαριστώ τον Πίτρο Πονταλή. Έχουμε ε, επτά ψηφίσματα και τώρα ε, ε, εφόσον έληξε